Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Άρχεται η συνεδρία. Και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπάτηση εκπροσώπου της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Υποθέσεις Ασφάλειας, που εκπροσωπείται σήμερα από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριο Στυλιανίδη. Καλώς ήρθατε. Για το θέμα, η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στην βορειοανατολική Συρία και οι επιπτώσεις της. Όπως ξέρετε, έχουμε ένα νέο σύστημα για τις μπλε κάρτες. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω συνέχεια πώς λειτουργεί. Ωστόσο, από τη μία μπορείτε να αξιοποιήσετε την παραδοσιακή μορφή αίτησης λόγου και από την άλλη ηλεκτρονικά. Δεν χρειάζεται να περιμένετε να περάσουμε στη φάση του catch the eye. Οπότε να περάσουμε απευθείας στη συζήτηση για το θέμα αυτό και να δώσω το λόγο και πάλι στην εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την κυρία Τούτι Τουπουράινεν. Παρακαλώ ε, να μας παρουσιάσετε την άποψη του Συμβουλίου. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Η εισβολή των Τούρκων στη βορειοανατολική Συρία μοιάζει να έχει επιβραδυνθεί. Βλέπουμε ότι διάφοροι διεθνείς παράγοντες έπαιξαν ρόλο για να υπάρξει αυτή η επιβράδυνση. Είπαμε είδαμε πολλέ ε, διπλωματικές προσπάθειες για να αποκλιμακωθεί η ένταση. Πρώτα απ' όλο ο αντιπρόεδρο Πεν και ο υπουργός εσωτερικών Πόμπεο που ε, διαπραγματεύτηκαν μία προσωρινή κατάπτωση του πυρός. Επίση υπάρχει ένα μνημόνιο που χθε υπεγράφει μεταξύ του πρόεδρου Πούτιν και του πρόεδρου Έρντοαν στο Σότσι. Η είπατε ήταν στο κοινοβούλιο την πρώτη μέρα τη επίθεση, και αμέσω κατέστησε σαφή την πρόθεσή μα. Η Τουρκία πρέπει να σταματήσει αμέσω την επίθεση. Βεβαίω, οι ανησυχίε τη πρέπει να αντιμετωπιστούν, αλλά διπλωματικά, όχι μέσω στρατιωτική δράση, που το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να αποσταθροποιήσει περαιτέρω την περιοχή και να ε, επιφέρει περισσότερα δυνάρια για το συριακό πληθυσμό. Επιπλέον, θεωρούμε ότι οι ανθρωπιστικοί οργανισμοί δεν θα έπρεπε να σταματήσουν να βοηθούν. Και όσοι έχουν μετατοπιστεί ε, λόγω του φόβου των συγκρούσεων έχουν αρχίσει να επιστρέφουν. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχει καμία δικαιολογία για τις ε, περίπου 200 περιπτώσεις θανάτου αμάχων ούτε για το βομβαρδισμό εγκαταστάσεων ίδρυυση νοσοκομείων και ασθενοφόρων. Ανησυχούμε για την μοίρα των Κούρδων της Συρίας και για όλους τους αμάχους στην ε, περιοχή των εχθροπραξιών. Η μόνη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν οι προσδοκίε και να αναγνωρίσουμε τι θυσίε που έκαναν οι, Σύρι, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ε, στην καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους είναι να δημιουργηθεί μια Συρία δημοκρατική, χωρίς αποκλεισμούς που όλοι οι πολίτες να αναγνωρίζουν ως την πατρίδα τους. Δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στην ε, Συριακή κρίση. Αντίθετα, πρέπει να στηρίξουμε την πολιτική διαδικασία για να υπάρξει μια μόνιμη λύση για όλους τους εμπλεκομένους. Οπότε, πρέπει να στηρίξουμε τη Συντακτική Επιτροπή που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στη Γενέβη στα τέλη του μήνα, παρά τις πρόσφατες εξελίξεις. Ή ακριβώς λόγω των ε, προσφάτων εξελίξεων πρέπει επιτέλους η Επιτροπή αυτή να συνεδριάσει. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στον ειδικό απεσταλμένο Γκέρ Πέτερσεν των Ηνωμένων Εθνών και πιστεύουμε ότι μια σταδιακή πολιτική προσέγγιση μπορεί να εξευρεθεί. Μέσω αυτή τη Συντακτική Επιτροπή για ένα καινούριο Σύνταγμα μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό κύκλο εμπιστοσύνη και τελικά να υπάρξουν αναγκαίες αλλαγές για ένα ειρηνικό και σταθερό μέλλον για τη Συρία. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο οδός προς μια ε, ε, πολιτική μετάβαση μετά από διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολη. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε με τους ε, διεθνείς μας εταίρους και ναι, η Ρωσία και η Τουρκία θα συμμετάσχουν. Γιατί πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάται η Συρία. Η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η λογοδοσία πρέπει να υπάρξει για όλα τα εγκλήματα που έκαναν όλες οι πλευρές. Μέχρι και το Ιντλιμπ και την πρόσφατη επίθεση. Αυτό για να υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα και συμφιλίωση, την οποία όλοι επιθυμούμε για τη Συρία. Τώρα να στραφώ στην Τουρκία και τις ευθύνε της για την ε, παρούσα κατάσταση. Οι ανησυχίε για την ασφάλεια που έχει η Τουρκία στα σύνορα με τη Συρία δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν μέσω στρατιωτικών επεμβάσεων. Αυτή η επίθεση, αντίθετα, υπονομεύει την καταπολέμηση του Ισλαμικού κράτους και απειλεί την κοινή μας ασφάλεια. Η Τουρκία έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες διότι φιλοξενεί ε, πολλά εκατομμύρια προσφύγων εδώ και τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά η στρατιωτική της δράση κάνει μια ιδιαίτερα περίπλοκη κατάσταση, ακόμη δυσχερέστερη και προσθέτει σε μια περίπλοκη και δραματική κατάσταση περαιτέρω επιπλοκές. Γι' αυτό η ηγεσία της Ένωσης και οι Υπουργοί Εξωτερικών καταδίκασαν αυτή την εισβολή της Τουρκίας. Και γι' αυτό τα κράτη-μέλη αποφάσαν να ε, διακοπούν οι εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία. Αυτή η επέμβαση δεν πρέπει μόνο να σταματήσει προσωρινά, πρέπει να σταματήσει οριστικά. Επίσης το Συμβούλιο είπε ότι δεν θα δώσουμε βοήθεια αναπτυξιακή ή σταθεροποιητική εκεί που αγνοούνται τα δικαιώματα του τοπικού πληθυσμού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε σαφής και ενωμένη από την πρώτη μέρα αυτής της ε, εισβολής. Τα τρία θεσμικά όργανα έστειλαν ταυτόσιμα μηνύματα και ευχαριστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, συνεχιζόμενη στήριξή του για να υπάρξει μια πολιτική λύση υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ο Αντιπρόεδρος κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Ευχαριστώ. Αξιότιμε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας ενημερώσω για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Ασία. Μία κρίση που εκτελήχθηκε στις 9 Οκτωβρίου και έχει οδηγήσει σε σοβαρές απώλειες, εκτοπισμούς, καταστροφές ε, ε, των ε, κοσμικών υποδομών και γενικά μεγάλες μάχες σε ιδιαίτερα πυκνές σε πληθυσμό περιοχές. Έχουμε 200 άτομα που έχασαν τη ζωή τους και 200.000 αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν. Υπάρχουν πάνω από 150.000 άνθρωποι που ε, θα εκτοπιστούν ε, και θα προσταθούν σε αυτούς που, ε, τους 100.000 που ήδη ήταν σε προσωρινούς καταβλισμούς πριν την κρίση. θέλουμε να υπάρχει μια ασφαλής περιοχή για αυτούς τους ανθρώπους που πάσχουν από τους ε, αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Οι διεθνείς ΜΚΟ και οι διεθνείς οργανισμοί έπρεπε να εκενώσουν προσωπικό στο Ιράκ. Αφήστε με τώρα να υπογραμμίσω αυτό που μόλις είπε η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για, τις, ε, για τον θάνατο αθών πολιτών, ε, για την καταστροφή υποδομών ε, και για αυτούς που χάνουν τη ζωή τους επειδή θέλουν να βοηθήσουν τους υπόλοιπους. Υπάρχει βαθιά ανησυχία λόγω της θλιβερής κατάστασης την οποία βιώνουν οι υπάλληλοι στον τομέα της υγείας, στα νοσοκομεία. Υπήρξε, υπήρξαν σοβαρές καταστροφές λόγω των αεροπορικών βομβαρδισμών και υπήρχαν περιπτώσεις ε, που κόπηκε το ρεύμα, ούτε καν οι γεννήτρες δεν λειτουργήσαν λόγω των βαβαρισμών και υπήρξε στοχοποίηση ακόμα και των ε, ασθενοφόρων ε, και δεν μπόρεσε να ακοινωθεί κόσμος από την, γραμμή, την πρώτη γραμμή του πολέμου. Μάλιστα σκοτώθηκαν ή απήχθησαν και υπάλληλοι στον τομέα της υγείας. Και αυτό ε, προστίθεται στα όσα ήδη υπέφεραν οι άνθρωποι πριν την κρίση. Ε, κατά την εκένωση του διεθνούς προσωπικού ε, καταλαβαίνετε ότι ε, αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να κάνουμε, προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν δίνουμε την υποστήριξή μας ε, στο πεδίο ε, της μάχης. Αυτή τη στιγμή 38.000 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για αυτό το σκοπό και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όσο χρειάζεται. Όμως πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Είναι ύψης της σημασίας ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι άνθρωποι που δουλεύουν στον ανθρωπιστικό τομέα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς που τους χρειάζονται. Πρέπει επίσης να ληφθεί κάθε πρόνοια ώστε να ε, εξαλειφθεί ο κίνδυνος ε, για τα καραβάνια που μεταφέρουν την ανθρωπιστική βοήθεια και για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν πρέπει αυτοί να στοχοποιούνται. Επίσης, να σας θυμίσω η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την επιστροφή των προσφύγων στη Συρία. Πρέπει όλες οι επιστροφές να είναι ασφαλείς, εθελούσιες και αξιοπρεπείς, να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Ιδάλλως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι σε θέση να δώσει την απαραίτητη Το ίδιο γίνεται και με τις λεγόμενες ουδέτερες ζώνες που θέλει να καταστήσει η Τουρκία στα βόρεια τη Συρίας με σκοπό τελικά να στείλει εκεί πίσω τους πρόσφυγες. Να σα θυμίσω επίσης ε, και την πρόσφατη δήλωση των 28 Οποιαδήποτε προσπάθεια δημογραφικής αλλαγής είναι απαράδεκτη. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να παράσχει τη σταθεροποίηση και να δώσει αρρωγή σε περιοχές όπου αγνοούνται τα δικαιώματα του ντόπιου πληθυσμού. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει και υποστηρίξει τις προσπάθειες της Τουρκίας ε, να φιλοξενήσει εκατομμύρια πρόσφυγες ε, στην επικράτειά της. Όμως η στρατιωτική δράση της στη Βόρεια Συρία έχει επιδεινώσει ήδη την κατάσταση στο πεδίο. Χαίρομαι λοιπόν που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι ενωμένοι στην αντίδρασή τους έναντι της στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας. Δεν πρέπει όμως να δρανίσουμε. Η σύντομη εκεχηρία εν μέρη μόνο έγινε σεβαστή. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας σε κάθε μέσο που έχουμε για να σταματήσουμε τις εχθροπαραξίες, να σταματήσει αυτή η ανθρωπιστική τραγωδία και να δώσουμε κάθε αρρωγή ώστε να επανέλθει η κατάσταση στο φυσιολογικό και να βρεθεί μια πολιτική λύση υπό, ε, στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Ευχαριστούμε και Τώρα ξεκινάει η συζήτηση. Πρώτος έχει ζητήσει τον λόγο ο Μίχελ Γκάλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σώμα μας έχει ευρεία συνένεση. Καταδικάζουμε την εισβολή της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία που είναι κατά του διεθνούς δικαίου και θέλουμε να αποσυρθούν τα στρατεύματα από το συριακό έδαφος. Αλλά δεν είμαστε αφελείς. Ξέρουμε ότι χθε στο Σότσι υπήρξε μια συμφωνία και είναι λυπηρό ότι αυτή η συμπεριφορά έγινε δυνατή ε, μέσω της μονομερούς απόσυρσης των τουρκικών στρατευμάτων. Και αυτές οι ενέργειες απομακρύνουν ακόμη περισσότερο την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό στο ψήφισμά μας υπενθυμίζουμε ότι το Κοινοβούλιο το Μάρτιο ζήτησε την επίσημη διακοπή των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Απαιτούμε από το Συμβούλιο να εξετάσει ανάλογες και στοχευμένες κυρώσεις που δεν θα θίξουν την κοινωνία των πολιτών. Να μην, μας, ε, να μην έχουν ως επίπτωση να μην μπορούν οι Τούρκοι σπουδαστές να υποφελθούν από τον έρασμο. Πρέπει να δούμε ποια γεωργικά προϊόντα θα μπορούσαμε να σκεφτούμε. Εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις. Και ως ε, έσχατο βήμα θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την αναστολή της Τελωνιακής Ένωσης ο πληθυσμό ε, στη Βόρεια Συρία δεν θέλουν ούτε τη Ρωσία, ούτε την Τουρκία, ούτε το καθεστώ ε, Ασάντ. Και εκεί λοιπόν στο ψήφισμα καλούμε τα κράτη-μέλη για άλλη μια φορά να στραφούν προ το Συμβούλιο Ασφαλεία των ΗΠΑ για να υπάρξει ένα ψήφισμα που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο να δράσει με στοχευμένο τρόπο. Με τελικό στόχο να υπάρξει μια ζώνη ασφαλεία υπό την αιγύδα των ΗΠΑ για να ωφελήσει τον τοπικό πληθυσμό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κατυπήρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρασαν δύο εβδομάδες από την προηγούμενη Ολομέλεια και τη συζήτηση που κάναμε για την κρίση αυτή. Η δημιουργία μιας ζώνης ασφαλείας έχει γίνει τώρα μια ζώνη πολέμου λόγω της εισβολής της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία. Ποιοι έχουν νικήσει ο Ασάντο, Πούτιν, η Τουρκία, η Τουρκία, το Ιράν και το Άισις. Και οι τιμένοι βέβαια είναι οι πολίτες της βορειοανατολική συρία και η εξοπιστία βέβαια τη δύση. 218 άμαχοι έχουν σκοτωθεί. Πολλοί μαχητές επίσης, πάνω από 300 άμαχοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και προσπαθούν αυτή τη στιγμή να βρουν ε, ένα ασφαλές μέρος. Βλέπουμε ότι προλάβουν όλο και περισσότερο οι δυνάμεις του Ασάντ από το νότιο. Έχουμε επίσης ε, πολλούς μαχητές της ISIS, Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν φύγει από τις φυλακές. Νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο και με την δολοφονία μιας γυναίκας πολιτικού από την ομάδα των Κούρδων. Επίσης χρησιμοποιείται λευκός φόσφορος στα πυρομαχικά της Τουρκίας κατά των Κούρδων. Νομίζω ότι πραγματικά θα πρέπει να βρεθούν ενώπιν τη δικαιοσύνη ε, οι υπέτη των ιδεχθών αυτών πράξεων. Και οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι ε, κατά αυτόν τον τρόπο, μέσω της εκεχηρία, θα σωθούν ε, πάρα πολλέ ζωέ. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να συμβεί όμω κάτι τέτοιο. Χθε ε, είχαμε μια συμφωνία μεταξύ Ρωσία και Τουρκία, ε, όπου δίνεται αυτή τη στιγμή δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ζώνη 10 χιλιόμετρων στα σύνορα μεταξύ Τουρκία και Συρία. Πάλι όμω μιλάμε για πάρα πολλού εκτοπισμού και ουσιαστικά εδώ πέρα παραβιάζονται βασικέ αρχέ ε, του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για του πρόσφυγε. Εμεί έχουμε ζητήσει να υπάρχουν στοχευμένε κυρώσει κατά των αξιωματούχων τη Τουρκία, περιοριστικά μέτρα, καθώ επίση και ένα πλήρε εμπάργκο των οπλισμών και πέρα από οποιαδήποτε ιδεολογική πολιτική πεποίθηση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προστατεύσουμε αυτούς που υπέφεραν από την ISIS και πολέμησαν κατά της ISIS για τη δική μας την ασφάλεια. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πύρη. Ο κύριος Μαλίκ Ασμάνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η τουρκική στρατιωτική επέμβαση στη βορειοανατολική Συρία σίγουρα μας προκαλεί πάρα πολλέ ανησυχίες και οδηγεί σε ένα χάος στην όλη περιοχή. Αναφερόμαστε σε εκατοντάδες ε, θανάτους, ε, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που έχουν εκτοπιστεί, πάρα πολλέ εκτελέσεις που έχουν λάβει χώρα. Μαχητές ε, του ISIS έχουν διαφύγει από τι φυλακές εξαιτία τη επέλαση των Τούρκων και τη αποχώρηση των Αμερικανών και είναι πάρα πολύ πιθανό οι τρομοκράτε αυτοί να επιστρέψουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό αποτελεί απειλή στη δική μα την ασφάλεια, για του δικού μα του πολίτε, για τι δικέ μα τι κοινωνίε. Απευθυνόμενο λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέσαμε κάποια ερωτήματα, στείλαμε μια επιστολή στην κυρία Μογκερίνη, την οποία υποστήριξαν και προσυπέγραψαν 250 συνάδελφοι και του ευχαριστώ για αυτό. Και περασμένε εβδομάδε εξ ονόματο του Renew Europe, ερχόμενο και σε επαφή με τουρκικέ αρχέ, προσπάθησα να δώσω τέλο στη βία αυτή. Αλλά δεν καταφέραμε ουσιαστικά να πρωτοστατήσουμε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε ω απλοί παρατηρητέ να βλέπουμε να επεμβαίνουν άλλοι, η Ρωσία, το Ιράν, ο Ασάντ, γιατί καταλαβαίνετε ότι διακυβεύεται η ίδια δική μα ευρωπαϊκή ασφάλεια. Για την ομάδα Renew Europe ο ρόλο μα δεν σταματάει εδώ πέρα. Αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη μοναδική ευκαιρία να μιλήσει με μία ενιαία ξεκάθαρη φωνή. Μία ενιαία φωνή προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε προ την Τουρκία ότι δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση την υφιστάμενη κατάσταση. Και να καλέσουμε επίση την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει ήδη ισχυρά μέτρα από τώρα. Και ζητώ από του συναδέλφου μου να με υποστηρίξουν αυτή τη στιγμή, καλώντα επιτακτικά την ύπατη εκπρόσωπο να ξεκινήσει ένα διάλογο με τι τουρκικέ αρχέ προκειμένου να βρεθεί μια βιώσιμη λύση και προκειμένου ο Ερντογάν να τηρήσει την υπόσχεσή του να κρατήσει του μαχητέ τη Άιση στι ε, φυλακέ. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για περαιτέρω δράση. Για παράδειγμα, στοχευμένε οικονομικέ κυρώσει. Θα πρέπει και το ενδεχόμενο αυτό να εξεταστεί. Α καταφέρουμε να συσπηρωθούμε, α δείξουμε ενότητα, α δώσουμε τέλο τώρα στη βία. Το χρωστάμε αυτό στου ανθρώπου που ζουν στην περιοχή αυτή, αλλά το χρωστάμε και του Ευρωπαίου πολίτε. Σα ευχαριστώ πολύ ε, παρακαλώ πολύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βγείτε από το περιθώριο και να λάβετε αυτή τη στιγμή δράση. Ευχαριστούμε κυρία Στρίκ. Ε, Αξιότιμε Πρόεδρε, ακριβώ πριν από δύο εβδομάδε ξεκίνησε μια σχεδιασμένη στρατιωτική επίθεση στη Βόρεια Συρία από την Τουρκία. Σε δύο εβδομάδε έχουν χάσει τη ζωή του πολλοί πολίτε. 200.000 ε, ε, Σύριοι χρειάστηκε να εκτοπιστούν από τα σπίτια του και υπάρχουν 70.000 ε, παιδιά που χρειάζονται καταφύγιο και υπάρχει, υπήρξε ανάγκη ακόμα και ανθρωπιστικέ οργανώσει να φύγουν από τη χώρα. Πρόκειται για μια ανθρωπιστική τραγωδία η οποία δεν πρέπει να συνεχίσει με την απόσυρση των στρατευμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι, Σύριοι, οι άνθρωποι της Συρίας έμειναν χωρίς καμία άλλη επιλογή παρά μόνο να περιμένουν με την οποιαδήποτε λύση εφεύρει ο Ερντογάν. Ε, πρέπει <clears throat> να, ε, να, να παραδεχτούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν φαίνεται πιθανότητα αποκλιμάκωσης της κρίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να δράσει με, ως ε, προμηθέας. Πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να ε, εμποδίσουμε το να γίνει απέλαση των Σύριων πίσω στη Συρία, των προσφύγων. βλέπουμε ότι ήδη έχει επιβληθεί ένα εμπάργο κατά των όπλων και μια αναστολή των εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει επίσης να προστατεύσουμε τους πρόσφυγες, ε, προσπαθώντας να μιλήσουμε υπέρ ε, της επανεγκατάστασής τους. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Κάνουμε έκκληση για το προτινόμενο ψήφισμα, λοιπόν. Οι τρομοκράτες του ISIS επίσης ξέφυγαν, διέφυγαν από τα φυλακές και αυτή τη στιγμή υπεκφεύγουν και της ε, δίωξης. Θα πρέπει να επαναπατρίσουμε ε, στην Ευρώπη τους ανθρώπους που ήταν μαχητές του ISIS και είναι Ευρωπαίοι πολίτες και να φροντίσουμε τα παιδιά τους. Αυτό για να μειώσουμε τον κίνδυνο ασφαλείας και να εμποδίσουμε την θυματοποίηση των παιδιών ένας από τους ρόλους της εισβολής του Ερδογάν είναι να απελάσει τους Σύριους ε, στη χώρα τους. Όμως, ακόμα και αυτές που αποκαλούνται ασφαλείς ζώνες δεν τους προστατεύουν από τη βία και την ε, δίωξη. σύμφωνη με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην επιστρέψει ε, Σύριους ε, πρόσφυγες στην Τουρκία όσο υπάρχει κίνδυνος απέλασης. Η απέλαση επίσης σημαίνει δημογραφική αλλαγή στον πληθυσμό της Βόρειας Συρίας. Αυτό είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Οι Κούρδοι που πάλεψαν στο πλευρό μας θα χάνουν την αυτονομία τους. Ε, πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε ότι ε, εμείς ως Ευρώπη ότι τα δικαιώματά τους γίνονται σεβαστά. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε εκ των προτέρων. Ευχαριστούμε. Κύριος ε, Λάνης Πάτρικ Μπέρκ. Ε, λυπάμαι και εκπλήσωμαι ε, όταν δεν τηρείται η εκεχηρία. Εκατοντάδες άνθρωποι ε, έχασαν τη ζωή τους λόγω της επίθεσης των Τούρκων και προδόθηκε ο κουρδικός λαός, ο εμείς ε, ε, τους είχαμε σύμμαχούς μας και τώρα τη στιγμή της ανάγκης έμειναν μόνοι τους. Ακούσαμε τις λυπηρές δηλώσεις ε, του Ερτογάν. Ε, υπάρχουν διάφοροι ετούντες άσυλο που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη και εμείς μιλάμε για την αποσταθεροποίηση, όμως αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρο πως η τουρκική συμπεριφορά είναι κατά του δικαίου. Ως τώρα, με τη δράση της ε, άφησε ελεύθερο το πεδίο στους ακραίους ε, και τους, τρομοκρα... τους τρομοκράτες. Εμείς στην Ευρώπη λοιπόν είμαστε σε μεγάλο κίνδυνο. Θα πρέπει ε, να έχουμε στο μυαλό μας με το ότι το SDF αν είναι ένα από τα πιο ε, επικίνδυνα, ε, μία από τις πιο επικίνδυνες οργανώσεις και δεν πρέπει πραγματικά όλα αυτά να τα αφήσουμε να έρθουν στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε η κυρία Άννα Φωτίγκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολλά σφάλματα έχουν γίνει από τη διεθνή κοινότητα στη Συρία και ήδη αυτό από το 2011. Πρέπει λοιπόν ε, να θυμόμαστε τις βιότητες του καθεστώτος του Ασάντα, στο Χαλέπι, επίσης την παρουσία των Ιρανών της Ιρανικής Επανεστατικής Πολιτοφυλακής στο, στη Συρία, καθώς επίσης και τους Ρώσους μισθοφόρους που ήταν βέβαια παρόντες και στην Ανατολική Ουκρανία. Προφανώς μας ανησυχούν πάρα πολύ οι πρόσφατες αυτές τρίτες κατά σειρά στρατιωτικές επεμβάσεις της Τουρκία, στην βορειοανατολική Συρία. Θα ήθελα να αναφέρω τον ε, Γενικό Γραμματέα Στότελμπεργκ, ο οποίο έκανε μία δήλωση το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που ήταν ιδιαίτερα ισορροπημένη η δήλωση αυτή. Είπε ότι μολονότι η Τουρκία έχει θεμητέ ανησυχίε όσον αφορά τον τομέα τη ασφάλεια, παρόλα αυτά περιμένω ότι η χώρα αυτή θα αναλάβει δράση με συγκράτηση. Και όλοι αυτό τελικά περιμένουμε, να δείξει συγκράτηση, αυτοσυγκράτηση η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, κάποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για όλους τους φορείς και παράγοντες στην περιοχή αυτή και θα πρέπει εμείς να καταφέρουμε να βρούμε τα κατάλληλα μέσα, τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να σταθεροποιήσουμε την περιοχή αυτή και προκειμένου να καταφέρουμε έτσι να έχουμε μια κάποια επίδραση σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν τελικά να μειώσουν την ένταση στην περιοχή. Επόμενη ομιλήτριά μας, η κυρία Özlem Demirel. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι Κούρδοι ενώ έκαναν τη δική μας δουλειά τώρα εγκαταλείφθηκαν. Και είναι απαράδεκτες οι δηλώσεις του ε, Τραμπ που φέρτε σαν παιδί. Πολλοί πέθαναν, ε, πολλοί προσπαθούν να αποφύγουν την ε, επίθεση. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε μία χώρα να επιτίθεται σε κάποια άλλη. Η κυβέρνηση Ερντοάν έχει γεωστρατηγικούς στόχους και η λεγόμενη ζώνη ασφαλείας δεν είναι ζώνη ασφαλείας. Είναι μια προσπάθεια να αλλάξει η διαμόρφωση της Συρίας. Όλες οι παγκόσμιες δυνάμεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολούνται με τα δικά τους οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα και κάθονται στο πλάι και βλέπουν να γίνονται εγκλήματα πολέμου και να καταπατείται το διεθνές δίκαιο. Ούτε πραγματικά ένα αγνήσιο εμπάργο όπλων δεν έχει επιβληθεί. Όλοι γνωρίζουν ότι ο Ερντοάν δεν θα μπορούσε να συνεχίσει τον πόλεμο του αν η διεθνή κοινότητα μιλούσε με την ίδια γλώσσα και αν υπήρχαν ε, βαριές οικονομικές κυρώσεις. Αυτό απαιτούμε. Πραγματικό εμπάργο όπλων. Καμία οικονομική σχέση πλέον με το κόμμα του Ερντοάν. Να υπάρξουν σωστές δομές στη Ροζάβα. Πρέπει να υπάρξει μια ειρηνική λύση για την περιφέρεια, για τη Συρία και καμία, υπογραμμίζω καμία στρατιωτική λύση. Η Ροζάβα είναι το παράδειγμα. Τα παιδιά, οι Κούρδοι και οι Συριακέ Δημοκρατικέ Δυνάμει είναι προοδευτικέ δυνάμει. Πρέπει να τι στηρίξουμε. Και ακόμη και αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα δικά τη γεωστρατηγικά συμφέροντα, ο πληθυσμό, η δημοκρατία, η ειρήνη και η ισότητα ε, δικαιωμάτων πρέπει να είναι το μέλημά μα. Ραντακόφσκι, ο κύριος Μύροσλαβ Ραντακόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Καταδικάζω την στρατιωτική επίθεση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία χωρίς καμία εντολή των Ηνωμένων Εθνών έγινε αυτή η επέμβαση χωρίς ε, βεβαίως ε, την ε, έγκριση των Σύρων. Αυτή η τουρκική επίθεση πρέπει να αντιμετωπιστεί με σκληρά μέτρα. Οι επιπτώσεις αυτής της επιθετικότητας θα είναι ροές τρομοκρατών προς την Ευρώπη. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να παίζει τον πολιτικό της ρόλο, τότε πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρξουν κυρώσεις. Να, να αρθούν οι κυρώσεις προς τη Συρία. Να ξεκινήσουμε και πάλι διπλωματικές σχέσεις με τη Συρία. Και να κάνουμε κάθε διπλωματική προσπάθεια για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Χωρίς παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας. Εάν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, Πρέπει να καταδικάσουμε την παρουσία όλων των ξένων δυνάμεων στη Συρία. Και με αυτόν τον απλό τρόπο θα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χαλίτσικη. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας με το κουρδικό έθνος και ελπίζω να εγκρίνουμε το ψήφισμα για το θέμα αυτό αύριο. Οι Κούρδοι αγωνίστηκαν για τα συμφέροντα της Δύσης, για να ζούμε με ασφάλεια και για να πούμε ότι νικήσαμε το Ισλαμικό κράτος. Οι Κούρδοι τον νίξαν. Αγωνίστηκαν απελευθέρωσαν πολλές πόλεις της Συρίας. Οι Κούρδοι. Σήμερα λοιπόν τι προτείνουμε. Προτείνουμε μια τροπολογία στον προπολογισμό για να παγώσει η προταξιακή βοήθεια προς την Τουρκία. Στην παράγραφο 45. Και μπορεί αυτή να περάσει στο αποθηματικό. Όμω δεν πρέπει να μειώσουμε ε, την βοήθεια που δίνεται προ την τουρκική κοινωνία των πολιτών. Και η, τρο, η τροπολογία αυτή θα δείξει ακριβώς ότι καταδικάζουμε στι δολοφονίες των Κούρδων. Ο κύριος Πίτσουλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξετάζουμε σήμερα τις ε, επιπτώσεις της στρατιωτικής επέμβασης της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία και συζητάμε επίσης βέβαια και τη συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών που έχει εκπνεύσει αλλά έχουμε και μια νέα συμφωνία τώρα μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Τίθεται λοιπόν ένα αμφιβόλο η ίδια η εδαφική ακαιρεότητα της Συρίας. Από ό,τι φαίνεται η συμφωνία αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεχθή και δεν θα πρέπει να γίνει αποδεχθή. Τι γίνεται όμω για του Κούρδου, του μαχητέ, οι οποίοι πραγματικά συνέβαλαν προκειμένου να καταπολεμήσουμε το Ισλαμικό κράτο. Τι θα γίνει με του Κούρδου μαχητέ εκείνου, του οποίου δεν θέλουν να δεχθούν και του οποίου δεν θέλουν να αναλάβουν οι δυτικέ χώρε. Και τι θα γίνει με τον τοπικό πληθυσμό που δεν περιλαμβάνεται καν σε αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι ο βασικός μα στόχος θα πρέπει να είναι η εκεχηρία, η κατάπαυση του πυρός για όλε τι εμπόλεμε εχθροπραξίε και δεν θα πρέπει εμεί να είμαστε απλώ εξωτερικοί παρατηρητέ. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν τι κυρώσει καθώς επίσης και την απαγόρευση εξαγωγή όπλων και να προωθήσουμε όλες τις δυνατές οικονομικές κυρώσεις. Πώς μπορεί να πάρει όμως στρατηγικές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Συρία όταν η ίδια δεν κατάφερε να πάρει τις αποφάσεις αυτές που ήταν τόσο αναγκαίες στο παρελθόν όταν δεν είχαμε για παράδειγμα ομοφωνία για σημαντικότατα ζητήματα όπως η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Ευχαριστώ η κυρία Χίλτε Βάουτμαντς. Πρόεδρε, συνάδελφοι, ο Ερδογάν θέλει πραγματικά να μας ε, κλονίσει. Το 2016 ε, ορίσαμε μια πολιτική και ε, στην ουσία του δώσαμε χρήματα. Έχει τώρα τα κλειδιά στα χέρια του. Μπορεί να ανοίξει τις πύλες και να αφήσει τους μετανάστες να φύγουν. Ψάχνει μια ασφαλή ζώνη. Αυτό λέει, αυτό ισχυρίζεται. Αυτό που εμείς όμως ε, ξέρουμε είναι ότι θέλει απλώς να πατάξει τους Κούρδους. Τι κάνει λοιπόν η Ευρώπη, αναρωτιέται ο κόσμος, για να σταματήσει αυτό η άθλια σύραξη. Η Ευρώπη απλώς ε, κοιτάζει απαθής. Ο Πούτιν υποστηρίζει το δικτατορικό καθεστώς του Ασάντ και οι Αμερικανοί απλώς ε, φεύγουν. Η Ευρώπη ε, κοιτάει απλώς ε, και αυτό επιδεινώνει την κατάσταση. Εμείς είμαστε απλοί παρατηρητές εμείς όμως είμαστε αυτοί που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα βάρη αυτής της διαδικασίας, ε, τους πρόσφυγες, τους ε, ριζοσπαστικοποιημένους ε, μαχητές που θα φύγουν και θα διαδοθούν σε όλο τον κόσμο. Πρέπει πραγματικά να διασφαλίσουμε η ασφαλή ζωή, ζώνη να καλύπτεται από τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό θέλουμε. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει τη δική της πολιτική ασφαλείας δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε συνεχώς από τους Αμερικανούς και τους Ρώσους. Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι πάνω από 700 παιδιά ε, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ευρωπαϊκά στρατόπεδα ε, των μαχητών ε, θα πρέπει να φροντίσουμε ότι δεν θα υποφέρουν λόγω των αμαρτιών των γονέων τους. Πρέπει να έχουμε την δική μας πολιτική. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σερκέη Λαγκοντίνσκι. Δύο γκριζομάλιδες ε, γυραιοί κύριοι συναντήθηκαν ε, στην Μόσχα και αποφάσισαν ε, να χωρίσουν μία περιοχή. Αυτό το έκαναν γιατί εμείς αποτύχαμε, γιατί οι θεσμοί μας απέτυχαν, γιατί το Κοινοβούλιο δεν εξυπηρετεί το σκοπό του ούτε και το Συμβούλιο, ούτε και η Κομισιόν. Ε, πού είναι τα μέτρα για τη συνολικό εμπάργο των όπλων, ε, πού είναι οι κυρώσεις για τις οποίες μιλάμε. Δεν μπορέσαμε να αναλάβουμε ευθύνη για αυτή την περιοχή και κάποιος άλλος την ανέλαβε. Δεν είναι όμως αργά. Πραγματικά μπορούμε ακόμα να γίνουμε ένας πολιτικός ε, να έχουμε ομόφωνες αποφάσεις στην εξωτερική πολιτική, να επενδύσουμε σε περισσότερη διπλωματία, σε περισσότερες πολιτικές εξωτερικής πολιτικής. Έχουμε τα επόμενα χρόνια για να το κάνουμε. Όχι για αυτούς τους ανθρώπους δυστυχώς και λυπόμαστε. Όμως τα επόμενα πέντε χρόνια έχουμε τη δυνατότητα να εμποδίζουμε τους γκριζομάλιδες να αναλαμβάνουν την ε, μοίρα των ανθρώπων στα χέρια τους. Έχουμε περισσότερους ανθρώπους, θέλουμε περισσότερες γυναίκες να αποφασίζουν για το μέλλον του κόσμου. Και κάτι άλλο να πω. Υπάρχει μία συνένεση εδώ, όπως είπε και ο κύριος Γκάλερ. Υπάρχουν πολλές πολιτικές δυνάμεις ε, ε, που ε, ψηφίζουν σκληρά ψηφίσματα. Αυτό όμως το κάνουν για διάφορους πολιτικούς λόγους. Θα σας πω εγώ γιατί ψηφίζουμε αυτά τα σκληρά λόγια. Θέλουμε να διασφαλίσουμε το ευρωπαϊκό μέλλον της Τουρκίας. Για να το διασφαλίσουμε λοιπόν πρέπει να δαμάσουμε τον υπεριαλισμό της κυβέρνησης της Τουρκίας, ε, τον, ε, την στρατιωτική στάση την ε, στάση που αντιτίθεται στον ανθρωπισμό γιατί υπάρχουν πολίτες, καλλιτέχνες, άνθρωποι στη φυλακή. Για αυτούς αξίζει να δώσουμε τη μάχη. Αυτοί θέλουν να ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα για να μην υπάρχει αυτό το μέλλον στην Τουρκία. Και το λέμε ξεκάθαρα, ψηφίζουμε αυτά τα σκληρά λόγια για να επιτρέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν ένα μέλλον στη δημοκρατία και στην Ευρώπη. Κατά το Ερντογάν, αλλά υπέρ της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ιβάν Ντάβιτ. Κοιτάξτε, θα ήμουν ε, απρόθυμος να υπερψηφίσω το ψήφισμα όπως είναι διατυπωμένο αυτή τη στιγμή. Διότι τα πιο κατηγορηματικά στοιχεία του ψηφίσματος διαγράφηκαν και προσθέθησαν φράσεις με τις οποίες δεν μπορώ να συμφωνήσω. Νομίζω ότι κάνουμε πολύ λίγα πράγματα και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Διότι οι Κούρδοι υφίστανται τις συνέπειες. Οι Κούρδοι που έκαναν τις θυσίες προηγουμένως. Και το χειρότερο είναι ότι όλα αυτά που γίνονται βασίζονται στη στην συμφωνία που συνήφθη στα Άδανα στη Συρία, όπου η Συρία και η Τουρκία απεκάλυψαν τους Κούρδους τρομοκράτες. Ενώ οι Κούρδοι νίκησαν το Ισλαμικό κράτος. Αυτοί αγωνίστηκαν για μας. Και η Ευρώπη, για άλλη μια φορά, δείχνει την αδυναμία της και την απροθυμία της να δράσει. Μόνο ένας οικονομικός αποκλεισμός μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ασίτα Κάνκο. Καλημέρα σας. Όταν ήμουν παιδί, αν κάποιος έλεγε ότι θα έρθουν οι Αμερικανοί να μας σώσουν, τους πίστευα γιατί είχα δει τις αμερικανικές ταινίες. Αν ήμουν ακόμη παιδί και κάποιο μου έλεγε τώρα, περίμενε, η Ευρώπη θα έρθει να σε σώσει. Μάλλον θα προσπαθούσα κάποια άλλη λύση να βρω. Διότι η διπλωματία μπορεί να φαίνεται ωραίο και ισχυρό μέσο. <clears throat> Αλλά αυτό μπορεί να έχει αποτελεσματικότητα μόνο αν υπάρχει καλή θέληση από την άλλη πλευρά. Στην ουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς μιλάει. Ενώ ορισμένοι μάχονται για την ελευθερία. Θα πρέπει να σταματήσουν οι εξαγωγέ όπλων στην Τουρκία και να επιβληθούν οικονομικέ κυρώσει. Θα πρέπει να υπάρξει απαγόρευση πτήσεων στη Βόρεια Συρία και να συνεχιστούν οι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει με συμμετοχή εκπροσώπων των Κούρδων. Πρέπει να διακοπεί η προενταξιακή βοήθεια ενώ θα εγγυόμεθα ανθρωπιστική βοήθεια για τους μετατοπιστέντες, για αυτούς που κινδυνεύουν. Δεν είναι δυνατόν να αποφεύγουμε τις ευθύνες μας. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει περισσότερα και να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις γυναίκες που υφίστανται τα πάνδυνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νικολάη Βίλουμσεν. Αμίνα Ματίνια. Είναι μια γυναίκα 73 ετών που σκοτώθηκε από χειροβομβίδες. Όπως και ο Ασίμ Χουσέιν, 11 ετών. Όπως η Μπρέιμα Αρμούσα, 3 ετών που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι. Ο Χουσέιν Άλι Κλάιν, 2 ετών παιδί, που έχει σοβαρά εγκάβματα. Ο κατάλογος ε, των θυμάτων είναι μακροσκελής των θυμάτων της εισβολής ε, του Ερντοάν στη βορειοανατολική Συρία. Η τουρκική στρατιωτική επέμβαση, οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι διάφορες ε, σύμμαχες πολιτοφυλακές εξετέλεσαν αμάχους, χρησιμοποίησαν χημικά όπλα, κατέστρεψαν πόλεις. Είδαμε ότι ο Τραμπ με την πολιτική του επέτρεψε να όλα αυτά. Εγκατέλειψε τους ε, συμμάχους μας, τους Κούρδους είδαμε ότι ο Ερντογάν συνεχίζει να διαπράττει τα εγκλήματά του, ενώ η Ένωση κοιτάζει απαθής. Και χθε τι είδαμε, ο Πούτιν και ο Ερντογάν συναντήθηκαν στο Σότσι και τα βρήκανε. Πώς θέλουν να μοιραστούν τα λάφυρα. Ενώ εμείς καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε. Η Τουρκία και η Ρωσία συνεχίζουν να βιάζουν την περιοχή και θέλουν να προχωρήσουν ακόμη περαιτέρω. Θέλουν να εισβάλλουν σε χριστιανικές ε, περιοχές της Βόρειας Συρίας. Αυτό είναι εθνοκάθαρση. Πρέπει να υπάρξουν κυρώσεις που θα επιφέρουν την κατάρρευση της τουρκικής οικονομίας και τη διακοπή της εισβολής. Μπορούμε να σταματήσουμε τον Ορντοάν αν έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους να δράσουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κωνσταντίνου. Κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια της προηγηθής ενημερώσεως σχετικά με τις τουρκικές επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία και με βάση τα διαλαμβανόμενα σε ειδησιογραφικές πληροφορίες διεθνών μέσων μαζικής επικοινωνίας, επιθυμώ να επισημάνω τα εξή. Η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας εναντίον των κουρδικών δυνάμεων προκάλεσε ήδη μαζικό εκτοπισμό πληθυσμού επίσης υπήρξαν ποικίλε αναφορές για αδιάκριτες επιθέσεις κατά αμάχων. εάν αυτό το στοιχείο επαληθευτεί συνεπάγεται πως αυτές οι επιθέσεις θα αποτελούν εγκλήματα πολέμου. αυτό το ενδεχόμενο μάλιστα τονίστηκε και στη δήλωση του αμερικανού υπουργού άμυνας έσπερ. οφείλω επίση να τονίσω τη χθεσινή δήλωση του james jeffrey του ειδικού απεσταλμένου του αμερικανού προέδρου για τη συρία ότι δεκάδες τζιχαντιστές του ισλαμικού κράτους αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την έναρξη της εισβολής του τουρκικού στρατού στη βορειοανατολική συρία. για τα δύο προαναφερθέντα στοιχεία οφείλουν τα όργανα της ενώσεως να επιδείξουν συστηματική ενάργεια στην αντιμετώπιση τους. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μακάλιστερ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι συνάδελφοι, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας ε, στη Βόρεια Συρία είναι ένα γεγονός που μας καταρακώνει, είναι μια σύρεξη λυπηρή. Θα έχει στρατιωτικές επιπτώσεις, αλλά προκαλεί και ε, προβλήματα δεινά στον τόπιο πληθυσμό και ε, απελευθερώνει τον Ισλαμικό, την Ισλαμική τρομοκρατία το ΕΛΚ, το ΑΛΔΕ, όλοι οι συνάδελφοι το ανέφεραν σήμερα το πρωί. Θα ήθελα συνάδελφοι να σας ενημερώσω, ότι ως πρόεδρος της ΑΦΕΤ μαζί με τους επιτρόπους ε, της Επιτροπής ε, Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου ε, εξεδώσαμε κοινή δήλωση για το θέμα αυτό. Θεωρήσαμε ότι η εγκατάλειψη των κουρδικών δυνάμεων και των συριακών δημοκρατικών δυνάμεων δυνάμεων ε, ήταν ε, απαράδεκτη καθώς μας βοήθησαν κατά του ISIS στη Συρία. Ε, φαίνεται ότι το γεγονός της απόσυρσης των στρατευμάτων των ΗΠΑ έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ζητάμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλους ε, τους, ε, και όλους ε, τους υπόλοιπους φορείς να αναλάβουν δράση έτσι ώστε να έχουμε μια ισχυρή και συνολική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την κρίση. Σας ζητώ λοιπόν να ληφθούν πρωτοβουλίες για να έχουμε διεθνή έλεγχο μια ζώνη αυσαλίας στη Συρία η οποία θα σταθεροποιήσει την περιοχή και θα ξαναδώσει τη δυνατότητα να ζήσουν οι πολίτες εκεί ασφαλείς. Ευχαριστώ.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 Πρώτα απ' όλα να μιλήσετε λίγο πιο αργά. Συγγνώμη για τη διακοπή. Σας παρακαλώ να μιλάτε λίγο αργότερα, λίγο πιο σιγά για τους διερμηνείς. Εντάξει. Ευχαριστώ. Όπως είπε το Συμβούλιο και είναι και θέση της ομάδας μου, η στρατιωτική επέμβαση των Τούρκων στη Συρία αποτελεί σαφή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επιπλέον, είναι από πολλέ απόψει απαράδεκτη. Αλλά πρώτα θέλω να πω ότι το διεθνέ δίκαιο πρέπει να είναι το πλαίσιο για όλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το χρησιμοποίησε για να υπάρξει ανοικοδόμηση και ειρήνη. Για να υπάρξει ένα νέο σύνταγμα. Καμία όμω από τι ανησυχίε για θέματα ασφάλεια που αναφέρει η Τουρκία δεν μπορεί να αιτιολογεί αυτή την εισβολή. Δεν είναι λύση. Είναι πρόλογο ε, των μετέπειτα προβλημάτων. Η Τουρκία είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Θα μπορούσε να ζητήσει την αλληλεγγύη των συμμάχων της. Δεν μπορεί να δρά εκτός του διεθνούς πλαισίου. Το γεγονός ότι φιλοξενεί πάρα πολλούς ε, Σύρους πρόσφυγες δεν σημαίνει ότι μπορεί να εισβάλλει στη χώρα τους. Και να εισβάλλει στην επικράτεια της άλλης ε, χώρας δεν μπορεί να βοηθήσει τη χώρα διότι έτσι ε, αλλάζει τις ισορροπίες από δημογραφικής και πολιτικής πλευράς. Και αυτό το κενό που δημιουργείται δεν ξέρουμε ποιος θα το ε, γεμίσει. Η μόνη δυνατότητα είναι να επιστρέψουν ε, θελοντικά στις αιστείες τους οι Σύριοι πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Κυρία Φονβίζε, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όταν εισέβαλε η Τουρκία, περίπου 7.000 παιδιά των μαχητών ISIS ζούσαν σε καταβλισμού στη Βόρεια Συρία. Ανάμεσα στα παιδιά αυτά, περίπου 700 ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Πολλά αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν και δεν γνωρίζουμε πλέον τη μοίρα τους που βρίσκονται. Δεν μπορούμε εμείς να εγκαταλείψουμε τα παιδιά αυτά, ούτε μπορούμε να τα τιμωρούμε για τα εγκλήματα των γονιών τους. Κανένα παιδί κατά των 10 δεν θα πρέπει να θεωρείται ποινικά υπεύθυνο σε κανένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνω έκκληση λοιπόν προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμμορφωθούν με τους εθνικούς, ευρωπαϊκούς αλλά και διεθνείς νόμους προκειμένου να επαναπατριστούν τα παιδιά αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτού είναι πολύ αργά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Για 1,5 λεπτό τώρα η κυρία Μπρικμό έχει το λόγο. Κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, κλείστε για μια στιγμή τα μάτια ακούγοντας την παρέμβασή μου. Έχετε παιδιά και το μεγάλο, παιδί, το μεγάλο σας παιδί που το αγαπάτε πάρα πολύ και το οποίο ζει στο Βέλγιο φεύγει για μία μάχη. Εσείς προσεύχεστε να επιστρέψει. Δεν επιστρέφει. Λείπει πολιτική βούληση. Τα παιδιά σας γεννιούνται λοιπόν στο περιβάλλον αυτό πολέμου, σε συνθήκες υποσυτισμού. Ο γιος σας αυτός πεθαίνει για μια μάχη την οποία δίνετε κι εσείς εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δίνετε μια μάχη στη συνέχεια προκειμένου τα παιδιά σας τα οποία δεν φταίνε τίποτα, δεν ευθύνονται για τον πόλεμο αυτό, τα υπόλοιπα παιδιά να καταφέρουν τουλάχιστον να επαναπατριστούν στην Ευρώπη. Ως βουλευτές λοιπόν, άντρε και γυναίκες έχουμε τώρα τη δυνατότητα αυτή να καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε τα παιδιά αυτά που είναι υπήκοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε να συντονίσουμε εμείς ω Ευρωπαϊκή Ένωση τη δράση αυτή επαναπατρισμού και να βασιστούμε επίσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση και τα δικαιώματα του παιδιού, την οποία καλούμε θα όλοι να τηρούμε. Σας ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό. Ο κύριος Μαριανή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο σε μια ανάρτησή μου στο Twitter έλεγα ότι σε τελευταία ανάλυση οι μόνοι που θα προστατεύσουν τους Κούρδους της Συρίας από τις απόπειρες εξάλληψης των Τούρκων είναι το καθεστώς Ασάντ. Μπορεί να σας κάνει εντύπωση η θέση μου αυτή, αλλά ήταν εντελώς προβλέψιμη. Εντελώς προβλέψιμη διότι πώς θα μπορούσαμε να αμφιβάλλουμε τελικά ότι θα εγκαταλείπονταν τελικά οι Κούρδοι από, αυτοί που τους, από αυτούς που τους υπόσχονταν ότι θα τους προστάτευαν. Πώς μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό ρητορικό από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίο είχε πει πολύ καιρό πριν τι εκλογέ ότι θα πέσει ρόλο στου Τούρκου στρατιώτε από τη Συρία για ποιο λόγο να μας εκπλήσει αυτή τη στιγμή η τουρκική παρέμβαση στη Σύρια που ήταν και αυτή τελώ προβλέψιμη και προφανώς αυτή τη στιγμή δεν υπερασπίζουμε την Τουρκία, καταδικάζω απερίφραστα την εισβολή τους, αλλά ουσιαστικά ποιο κράτος θα δεχόταν ποτέ να έχει στα σύνορά του τρομοκρατικέ τρομοκρατικές ομάδες που κάνουν συνεχώς επιθέσεις ε, στην Τουρκία. Τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή, διεθνέ δίκαιο, να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την κυριαρχία και κεραιότητα της Συρίας στο σύνολο της επικράτειας και να καταφέρουμε να προωθήσουμε τη συμφιλίωση και την ειρήνευση οι κυρώσεις αυτή τη στιγμή που βαρύνουν την Συρία όσον αφορά το νεατρικό εξοπλισμό ουσιαστικά επιδεινώνουν την κατάσταση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είχαμε ένα πολύ πιο στρατηγικό όραμα ως Ευρωπαϊκή Ένωση που να λαμβάνει υπόψη του τις ιδιαιτερότητες ε, της περιοχής αυτής. Είμαστε εξωτερικοί παρατηρητές, ε, συζητάμε, ψηφίζουμε ψηφίσματα, αλλά ποτέ δεν ήμασταν στο προσκήνιο πραγματικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει την πραγματική κατάσταση και να καταφέρει πραγματικά να έχει ένα στρατηγικό όραμα για την περιοχή αυτή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριο Στέρτστρο έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η τουρκική εισβολή στην Συρία αναμφίβολα είναι τραγωδία, αλλά ήταν ε, προβλέψιμη, διότι η Τουρκία έχει συμφέροντα στην περιοχή. Σοβαρά συμφέροντα και τα 3,5 εκατομμύρια Σύρων προσφύγων που φιλοξενεί η Τουρκία είναι σαφό, σαφές ότι πιέζει την Τουρκία και μέχρι σήμερα δεν καταλάβαμε τι συμβαίνει, μέχρι τώρα που συμβαίνει. Πρέπει φυσικά να ασκήσουμε πίεση στην Τουρκία για να σταματήσει αυτή την εισβολή, για να δημιουργηθούν ε, οι προστατευμένες ζώνες ασφαλείας. Ούτε την Τουρκία την ενδιαφέρει μία Παξ Πούτιν στην Συρία. Γιατί αυτό θα ωφελούσε μόνο τον ίδιο τον Πούτιν και το Ιράν. Η Ευρώπη απλώς ε, εκφράζει τη λύπη της, διότι δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Ενώ οι Αμερικανοί παντού θα συμβάλλουν ε, στη δημιουργία δεινών. Δεν υπάρχει λοιπόν ο αναγκαίος ρεαλισμός στην Ευρώπη. Οπότε δεν έχει κανένα μέλλον. Ο κύριος Γεωργίου, ένα λεπτό πάνω. και πολιτική ταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμάστε που θα φέρνετε μαζί με άλλους την άνοιξη στις αραβικές χώρες. Τώρα που ήρθε η βαριχημονιά, κλαίτε με κροκοδίλια δάκρυα επί των ερυπείων. Πριν από 8 χρόνια ξεκίνησε μια ξένη εισβολή σε βάρος της κυβέρνησης της Συρίας για να την ανατρέψει και για να διαμελήσει τη χώρα οι ηνωμένε πολιτείε τη Αμερική το νάτο η τουρκία χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μοναρχίε του κόλπου εξόπλισαν δια τη συριακή αντιπολίτευση τις ορδές των τζιχαντιστών και του ισλαμικού κράτου. τώρα με την ανοχή τη Ρωσία και τη Αμερική και με τι φραστικέ καταδίκες μόνο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αμολύθηκε ενός θηρίων ο ερντογάν για να πιει το αίμα και να ξανατσακίσει έναν πολύπαθον λαό τους Κούρδους. Κανένας δισταγμό, καμία ηθική αναστολή από κανέναν. Φτάνει να ξαναμοιραστεί η περιοχή, να πουληθούν όπλα, να βγει το πετρέλαιο και εν τέλει θεωρώ ότι ακούγονται όλα αυτά ως τραγελαφικά και μάλλον είμαστε τραγικοί. Τίποτα άλλο. Και ο κύριος Καστάλντο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πριν από ένα περίπου μήνα είχαμε την επέμβαση αυτή και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τις τραγικές επιπτώσεις και Amnesty International μας μιλάει γι' αυτό, ιδίως για τον άμαχο πληθυσμό και για πραγματικά εγκλήματα πολέμου γίνεται λόγος. Και πολλά κράτη-μέλη Δυστυχώ όχι όλα. Αποφάσισαν τότε να σταματήσουν τι εξαγωγέ όπλων προ την Άγκυρα. Αυτό όμω δεν αρκεί. Θα πρέπει εμεί να κλείσουμε οριστικά αυτή την φαρσοκομωδία τη ένταξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει επίση να μπλοκαριστεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να καταλήξει στι τσέπε του Ερντογάν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα λόγω τη συμφωνία αυτή και τη χρηματοδότηση προ την Τουρκία για την ανάσχεσή τη μεταναστευτική κρίση. Επίση, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που μπορούμε να έχουμε. Στοχευμένε οικονομικέ κυρώσει, μια συγκεκριμένη εμπορική πολιτική, να βάλουμε κατά συγκεκριμένων προτιμησιακών ε, προϊόντων κ.ο.κ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην εγκαταλείψουμε του Κούρδου για μία ακόμα φορά. Α μην το πράξουμε αυτό, τουλάχιστον εμεί οι Ευρωπαίοι. Ο κύριος Πασέσκου έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εισβολή της Τουρκίας στην βορειοανατολική Συρία έχει δύο πτυχές, θεωρώ. Μία πτυχή που έχει να κάνει με το τομέα της ασφάλειας διότι ουσιαστικά οι Τούρκοι θεωρούν ότι οι Κούρδοι μαχητές είναι τρομοκράτες, ενώ η άλλη πτυχή έχει να κάνει με τη μετανάστευση και έχει να κάνει και με τον ανθρωπιστικό τομέα. Οι επιπτώσεις της εισβολής αυτής είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Ο στρατός της Συρίας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει φτάσει στα βόρεια της χώρας. Αυτό ουσιαστικά εμπόδισε τα τουρκικά στρατεύματα από το να ελέγχουν το σύνολο της παραμεθορίου αναγκάστηκαν κατά αυτόν τον τρόπο να περιοριστούν σε μια ζώνη 120 χιλιόμετρων, σε σύνολο 400 χιλιόμετρων. Η επέμβαση όμως αυτή οδήγησε στον εκτοπισμό 160.000 Συρίων μέσα σε μερικές μονομέρες και 200 άμαχοι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτής της επέμβασης. Τέλος, η τουρκική αυτή επέμβαση επέτρεψε στον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να γίνει ξεχνικά ο θεματοφύλακας της μελλοντική ανεξαρτησίας και της μελλοντική εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Με άλλα λόγια, να καταφέρει να παγιώσει την επιρροή του στο σύνολο της Συρίας. Εμείς λέμε εδώ πέρα ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε τις εξαγωγές όπλων προς την Τουρκία, μα ένα πρόβλημα. Από τον Πούτιν θα αγοράσουν στο μέλλον τα όπλα τους. Διακόπτη πρόεδρος. αυτή η ζώνη ασφαλείας που θέλει να δημιουργήσει ο πρόεδρος Πούτιν θα πρέπει πραγματικά να μας απασχολήσει. Διακόπτη πρόεδρος, έδωξα μια κάποια ευελιξία στο χρόνο αγόρευσης, αλλά θα πρέπει να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Μιλήσατε το διπλάσιο χρόνο. Ας περάσουμε τώρα στον επόμενο μιλητή, είναι η κυρία Σάντος για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή ε, κανείς ε, ε, ε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η εισβολή στη Βόρεια Συρία είναι παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε εξαναγκασμένο εκτοπισμό των πολιτών, σε επιδείνωση της σύραξης και σε άνοιγμα της πόρτας στον ISIS. Δεν πρέπει να μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μίλησε για το εμπάργκο στα όπλα. Αυτό όμως δεν αρκεί. Πρέπει να καλύψουμε όλες τις ε, παραδόσεις, όλα τις παραδόσεις όπλων που αυτή τη στιγμή τρέχουν. Πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις έναντι όλων όσοι εμπλέκονται άμεσα στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να δράσουμε επί των οικονομικών συμφερόντων και να δείξουμε ξεκάθαρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκβιάζεται. Πρέπει να δώσουμε ανθρωπίνων ανθρωπιστική βοήθεια στις χώρες που δέχονται τους πρόσφυγες και δεν πρέπει να δεχόμαστε εξαναγκασμένοι ε, ο επανταμπατρισμό. Ε, θα πρέπει οι άνθρωποι να ε, έχουν μια εθελούσια επιστροφή με συνθήκες αξιοπρεπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν μπορεί να υποστηρίξει οποιαδήποτε διαχείριση της κατάστασης, της κοινωνικής κατάστασης με τρόπο εξαναγκαστικό οι ε, οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας ε, μαχήθηκαν στο πλευρό μας ε, κατά του ISIS και πρέπει εμείς να διατηρήσουμε την αλληλεγγύη μας προς αυτούς, γιατί αλλιώς θα έχουμε επιπτώσεις. Ε, για δύο λεπτά η κυρία Λουαζό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό που συμβαίνει στην νοτιο... στη βορειοανατολική Συρία αυτή τη στιγμή είναι μια τραγεγωδία οποία παίζεται το Σύριαλ εδώ και τόσα χρόνια. Η επίθεση της Τουρκίας, η οποία στοχεύει στους ε, Κούρδους, ε, στην ουσία ε, ανθρώπους οι οποίοι πάλεψαν κατά του ISIS στο πλευρό μας, μας οδηγεί σε μια κατάσταση εκτέλεσης πολιτικών ηγετών, όπως πριν Καλέφ. Υπάρχουν Ευρωπαίοι οι οποίοι κρατούνται και δεν υπάρχει επιτήρηση. αυτή αυτά τα δικαιώματα που εμείς χτίσαμε τώρα παραβιάζονται. Το ΝΑΤΟ ε, αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι ε, υπερασπίζεται τη δική μας ασφάλεια, όμως παρέλυσε και έχει πιαστεί εξαπίνης. Εμείς ε, δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ρωσία να ενισχύσει το ρόλο της στην Αγγίσσα Ανατολή. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι να αφήνουμε τους Αμερικάνους να μας θεωρούν αμεληταία ποσότητα στις επιλογές σας. Ε, γιατί όλα αυτά γίνονται ε, ρήμιν μας ε, και εναντίον μας. δεν είχαμε την στρατηγική αυτονομία που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ευρωπαϊκή άμυνα η οποία θα μας κάνει σεβαστούς, θα σέβεται την ασφάλειά μας γιατί αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα. για 1,5 λεπτό ο κύριος Ουρτασούν.